προτείνει μια ερμηνεία του παραρτήματος 16 του κανονισμού σε σχέση με τις ναι. κατευθυντήρες γραμμές για την ε, έγκριση της Κομισιόν. Θα βρείτε το κείμενο στην ιστοσελίδα της ε, Ολομέλειας. Αυτή η ερμηνεία θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί εάν μέχρι την αρχή τη επόμενη συνεδρία Ολομέλεια μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτέ δεν έχουν εγείρει αντίρρηση. Βάσει του άρθρου